Αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση. Η παρουσία των μελών επιδέχεται κάποια αύξηση. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης έχουν κατανεμηθεί. Έχετε καθόλου αντιρρήσεις.